Welcome back. Καλώς επιστρέψατε και παρακαλώ καθίστε. Χαίρομαι που είστε ακόμα εδώ. Ε, απομένει ακόμα λίγη ώρα. Κάναμε το διάλειμμα για καφέ και τώρα θα συνεχίσουμε και νομίζω ότι δεν έχουμε καθυστερήσει. Θα συνεχίσουμε μέχρι τις 5.30. όπου και θα ξεκινήσει το τελευταίο κομμάτι και το τελευταίο πάνελ. Βλέπω ότι είναι ήδη εδώ τα μέλη του πάνελ. Καλωσορίστε τον κύριο Βιβαρόφσκι, τον ε, ε, Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων και τον καθηγητή Πελεγκρίνη. τον κύριο Πελεγκρίνη, πρόεδρο του ε, Συμβουλίου Συνεργασίας της Ευρωπόλ. θα κάνουμε μια συζήτηση για τον εσωτερικό κανονισμό. Αυτό είναι το σημείο ουσιαστικά. Θα ασχοληθούμε με τις τροπολογίες που έχουμε υποβάλει όσον αφορά τον εσωτερικό κανονισμό. Για να σας δώσω το πλαίσιο δυνάμει του άρθρου 6 του εσωτερικού κανονισμού JPSG σε συμφωνία με τις συστάσεις της διάσκεψης αγορητών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 23 και 23. 23 και 24, 24 Απριλίου του 2017 στην Πρατισλάβα το GPSG θα πρέπει να αναθεωρεί τον εσωτερικό του κανονισμό δύο έτη μετά από την συνεδρίαση σύστασης του σε σώμα και να υποβάλει τα συμπεράσματα της αναθεώρησης αυτής στην Προεδρία της Διάσκεψης των Αγορετών των Κοινοβουλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βάσει αυτού η προθεσμία τροπολογιών ε, ορίστηκε στην τελευταία συνάντηση JPSG στο Βουκουρέστο Φεβρουάριο. Η προθεσμία είναι 4 Σεπτεμβρίου. Ήταν. Εντό τη προθεσμία υποβλήθηκαν 13 τροπολογίε από τι αντιπροσωπείε. Επιπλέον, ε, διάφορε τροπολογίε υποβλήθηκαν. Διάφορε ε, υποβλήθηκαν από συμπροέδρου ω αποτέλεσμα τη σκληρή δουλειά τη ομάδα εργασία για τη Δανία και τι συμμετοχέ των Βουλγαρικού, του Ρωμανικού, του Φιλανδικού και του Κροατικού Κοινοβουλίου στη διάρκεια της Προεδρίας τους με τη συμμετοχή, για τη συμμετοχή του Δανέζικου Κοινοβουλίου στο JPSG. Το JPSG επίσης έλαβε διάφορες γραπτές συμμετοχές που προτείνουν αλλαγές στον ιστορικό κανονισμό. Όλες οι τροπολογίες που έχουν ληφθεί και τα γραπτά σχόλια συμπεριλαμβάνεται στα έγγραφα της συνάντησης που έχουν δοθεί για την σημερινή μας συνεδρίαση. Υπάρχει ένα σύνολο τροπολογιών για τη συμμετοχή του Δανικού Κοινοβουλίου. Ξέρετε πώς έχουν τα πράγματα με τη Δανία. Η Δανία δεν συμμετέχει έχει διαφορετικές ε, συνθήκες ε, ε, στην συνθήκη της Λισαβόνας και διαπραγματεύτηκε της δική της ιδιαίτερη συμμετοχή στην στο ομάδα ελέγχου της Ευρωπόλου. Οπότε το πώς θα οργανωθούμε για να ασχοληθούμε με αυτές τις τροπολογίες τώρα προτείνω το εξής η Τριάδα Προεδριών συμφώνησε μια διαδικασία για τη συζήτησή μας και την έγκριση των τροπολογιών. Δύο επιλογές έχουμε. Σε περίπτωση τροπολογίας που υιοθετείται με συνένεση, το αποτέλεσμα θα είναι αλλαγή στον εσωτερικό κανονισμό. Σε περίπτωση δεύτερον μη συνένεσης σε μια τροπολογία, η τροπολογία δεν εγκρίνεται και διατηρείται στον ιστορικό κανονισμό το εν λόγω άρθρο όπως έχει αυτή τη στιγμή. Διατηρείται δηλαδή το status quo του ιστορικού κανονισμού. Και στις δύο περιπτώσεις, ε, κατά την άποψή μας, η συζήτηση Δευτέρας και Τρίτης θα είναι η τελική συζήτηση της διαδικασίας αναθεώρησης του εσωτερικού κανόνα του κανόνων για την αναθεώρηση του εστερικού κανονισμού. Προτείνω λοιπόν να ξεκινήσουμε με το πρώτο θέμα που έχουμε για τη συζήτησή μας. Ξεκινάμε με το σύνολο τροπολογιών για τη συμμετοχή του Δανικού Κοινοβουλίου στο JPSG. Ευχαριστούμε την προσοχή των αντιπροσωπιών σε αυτό στην κοινή μα επιστολή. Το σύνολο αυτών τροπολογιών επίση αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα IPEX όπω ονομάζεται. Το σύνολο αυτών τροπολογιών προτάθηκε από την ομάδα εργασία για τη συμμετοχή τη Δανία που αποτελείται από το την Τριάδα Προεδριών και το Δανικό, Δανέζικο Κοινοβούλιο. Στη συνέχεια υποβλήθηκαν, υποβλήθηκαν στο JPSG από του συμπρόεδρου τη ε, συνέδρια αυτή. Εμεί, ω συμπροέδροι προτείνουμε στις αντιπροσωπείες ε, να εγκρίνουν το σύνολο αυτό τροπολογιών ε, του εσωτερικού κανονισμού για τη συμμετοχή του Δανέζικου Κοινοβουλίου στο JPSG. Σύμφωνα με τις τροπολογίες του Κοινοβούλιο της Δανίας θα γίνει μέλος με περιορισμένα δικαιώματα στο JPSG αντί για το σημερινό του καθεστώς παρατηρητή. Θα προσθεθεί ένα πρωτόκολλο στον εσωτερικό κανονισμό. Σε αυτό το πρωτόκολλο θα ορίζονται οι προϋποθέσεις συμμετοχής του Δανέζικου Κοινοβουλίου για τους σκοπούς αυτούς. Το Δανέζικο Κοινοβούλιο δεν θα συμμετέχει στην διαδικασία λήψης αποφάσεων, αλλά η θέση του θα καταγράφεται. Θα μπαίνει στα πρακτικά δηλαδή. Οι συνεδριάσεις του JPSG δεν θα λαμβάνουν χώρα στη Δανία όταν η Δανία θα έχει την ε, Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Δανία δεν θα ορίζει τον εκπρόσωπο JPSG στο Διοικητικό Συμβουλίο της Ευρωπόλ. Αυτή είναι η θέση που εγκρίθηκε από όλους μας ε, τους συμπροέδρους ως αποτέλεσμα των εργασιών που προηγήθηκαν μέχρι στιγμής. Τώρα, για να εξηγήσει με την θέση του Δανέζικου Κοινοβουλίου επί του θέματος. Θα δώσουμε δύο λεπτά χρόνο αγόρευσης στον εκπρόσωπο του Δανέζικου Κοινοβουλίου, τον κύριο Ράσμους Νόρτβεστ, επικεφαλής της αντιπροσωπείας του Δανέζικου Κοινοβουλίου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ την Τρόικα, του συμπροεδρούς για τη δουλειά που έχουμε κάνει τα τελευταία δύο χρόνια. Ήταν δύσκολο να βρεθεί μια καλή λύση για να μπορέσει να έρθει και να εκπροσωπηθεί εδώ και το Κοινοβούλιο της Δανίας. Έχουμε κάνει καλή δουλειά όμως και η λύση αυτή τελικά είναι κάτι το οποίο όλοι θεωρούμε καλό και μπορούμε να συμμετέχουμε πλήρως ε, στις εργασίες της ομάδας. Θα ήθελα ιδιαίτερως να ευχαριστήσω το προσωπικό της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καθώς μας βοήθησαν να βρεθεί μια λύση η οποία θα επιτρεπόταν και από τον κανονισμό αλλά θα ανταποκρινόταν και στις επιθυμίες του Κοινοβουλίου της Δανίας για να μπορέσουμε να εργαστούμε εδώ. Οπότε είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι με τη λύση αυτή και ελπίζω και τα υπόλοιπα κοινοβούλια και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να στηρίξουν αυτή την αλλαγή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος... Σας ευχαριστώ κύριε Νόρτκριστ για την παρουσίαση αυτή. Τώρα βλέπω. Θέλει κάποιον λόγο. Έχει κάποια αντίρρηση. για το αποτέλεσμα της εργασίας. Ναι, παρακαλώ. Τι είστε, από την Πολωνία. Έχω μία αμφιβολία, γιατί δεν κατάλαβα καλά. Όταν θα ασκεί την Προεδρία η Δανία, την εκπεριτροπή Προεδρία της Ένωσης, ποιος θα ε, λάβει τη θέση της Δανίας στην τριάδα της Προεδρίας, στην Τρόικα των Προεδριών ε, ως και στη Europol. Γιατί εκπρόσωπος της 30ης Προεδρίας συμμετέχει ε, σε εργασίες της Europol. Η Τριάδα θα γίνει διάδα γιατί δεν θα συμμετέχει η Δανία. Πώς θα ρυθμίσουμε αυτό το θέμα της συμμετοχής της ε, στη Europol στα πλαίσια της Τριάδας Προεδριών. Κοιτάξτε, η διάταξη λέει ότι το προηγούμενο κράτος μέλος που, ε, το κράτος μέλος, που ακολουθεί στην εναλλασσόμενη Προεδρία θα αναλάβει και θα μπει στην Τρόικα για το σκοπό αυτό. Αυτό λόγω της ιδιαιτερότητας ε, της ε, ένταξης της ε, Δανίας. Οπότε θα είναι το επόμενο κράτος μέλος στην εναλλασσόμενη Προεδρία. Αυτό το οποίο ε, θα μπει στην Τρόικα. Αυτό θα γίνει. Αν δεν υπάρχουν άλλα σχόλια ή αντιρρήσεις, που μάλλον δεν υπάρχουν, τότε εγκρίνουμε αυτή την αλλαγή στον ε, κανονισμό ομόφωνα. Συμφωνείτε. Ωραία. Να σας ανακοινώσω. Ο κανονισμός θα τροποποιηθεί σύμφωνα με την απόφαση αυτή και η αλλαγή θα ισχύσει ε, από σήμερα ήδη, από τώρα. Εγκρίθηκε. Θα δώσω τον λόγο τώρα στην Σύμπροεδρο που θα προεδρεύσει στην υπόλοιπη συζήτηση και αφορά την αλλαγή του κανονισμού. Σας ευχαριστώ. Προτείνω τώρα να εξετάσουμε τις ε, προτάσεις για αλλαγές από τις αντιπροσωπείες. Ε, δύο λεπτά ο χρόνος ομιλίας. Λοιπόν, θα ακούσουμε τώρα τις ε, εξής προτάσεις. Πρώτα, την αντιπροσωπεία από τις ε, κάτω χώρες, κυρία Μόνικα Ντεμπούλ. Τροπολογία 158. Αγαπητοί συνάδελφοι, σας ευχαριστώ που έχουμε την δυνατότητα να υποβάλουμε τέτοιες ε, τροπολογίες, ε, κάτι το οποίο θα κάνουμε. Εμείς ε, θέλουμε να επιτύχουμε τέσσερις στόχους, δηλαδή να επιτύχουμε την διαφάνεια, να λειτουργούμε εγκαίρως, να υπάρχει συνέχεια, συνένεση και ουδετερότητα στην εκπροσώπηση. Τα θέματα των τροπολογιών αφορούν την έγκαιρη διάθεση των εγγράφων πριν από κάθε συνεδρίασή μας. Καθώς επίσης και την εισαγωγή την μιας απέτησης οι συμπρόεδροι να ε, εκθέτουν τους λόγους για τους οποίους απορρίπτουν αιτήματα. Θα εισαχθεί έτσι μια μέγιστη προθεσμία απάντησης από την Europol σε γραπτές ερωτήσεις γιατί γιατί θα έχουμε ήδη ε, διασφαλίσει την ε, έγκαιρη μετάδοση της απάντησης εντός 6 εβδομάδων. Και βεβαίω η Ολλανδική Αντιπροσωπεία προτείνει ή αντιπρόσωπος να έχει μια θητεία 18 μηνών. Θα πρέπει να ε, ορίζεται συνενετικά, αλλιώς με απλή πλειοψηφία και επιπλέον προτείνουμε η εκπρόσωπος να μην είναι από κάποιο κράτος μέλος της Τρόικας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και μετά από την Γερμανική Βουλή η κυρία Σουζάνε Μίταγκ. Τροπολογία 2. Mhm. Äh, Αγαπητοί συναδελφοί, κατά την απόψη μας ε, η πρακτική έχει δείξει ότι για να έχουμε πιο αποτελεσματικό έλεγχο και αποτελεσματικότερη εργασία στην ε, τροπολογία 2 ε, το ζήτημα είναι ότι μιλάμε για ένα σημαντικό κοινοβουλευτικό εργαλείο το οποίο προβλέπει έναν οργανισμό που θα πρέπει να έχει τη διάθεσή του επαρκής πληροφορίας για να κάνει εκτενώς τον έλεγχο. Ούτω ώστε όλα τα μέλη τη Επιτροπή να λαμβάνουν τι πληροφορίε και να μπορούν να τι χρησιμοποιήσουν στη δουλειά του, προτείνουμε στο 4.2 του εσωτερικού κανονισμού η διαβίβαση των ερωτήσεων και απαντήσεων να αποστέλλεται σε όλα τα μέλη της Επιτροπής και να δημοσιεύονται τα στοιχεία αυτά δεδομένων των νέων τεχνολογιών θα πρέπει αυτό να γίνεται πολύ εύκολα. Thank Σας ευχαριστώ. Τώρα, από την Τσεχική Βουλή, ο κύριος Γιαρόσλαφ Πετσό θα μας παρουσιάσει τις τροπολογίες 3 και 7, προτάσεις της Τσεχικής Βουλής. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Εγώ θα σας παρουσιάσω τις τροπολογίες της Τσεχικής Βουλής. Ήδη έχουμε παρουσιάσει την ιδέα αυτών των τροπολογιών στην συνεδρίαση του Βουκουρεστίου. Θεωρούμε ότι είναι σωστό και δίκαιο ε, εκπρόσωπός μας στην μεικτή ομάδα κοινοβουλευτικού ελέγχου να έχει την ίδια θητεία με την Προεδρία, ώστε να προλάβουν όλα τα κράτη-μέλη να διεκδικήσουν αυτή τη θέση του εκπροσώπου. Και σε ό,τι αφορά τη συνέχεια, είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί συνέχεια και στην υποβολή των εκθέσεων από τους ε, εκπροσώπους. Μέχρι στιγμής ήταν μονοσέλιδες οι εκθέσεις. Δεν ήταν και πολύ χρήσιμες. Βέβαια, αυτό επαφείται στη διακριτική ευχαίρεια του εκπροσώπου. Αλλά είναι σημαντικό να είναι πιο εκτενείς και πιο ενημερωτικές οι εκθέσεις. Επίσης, ό,τι αφορά τη δεύτερη τροπολογία, καλό θα ήταν να αλλάξει ο τρόπος ψηφοφορίας. Βέβαια, η ομοφωνία είναι το ζητούμενο και προτιμότερο, αλλά θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε και με έναν τρόπο ψηφοφορίας ε, που υιοθετείται αυτή τη στιγμή από την ΚΟΖΑΚ. Αλλά αν δεν μπορούμε να καταλήξουμε σε ομοφωνία, σχέση η ενισχυμένη πλειοψηφία. Θα μπορούσαμε να δεχτούμε και αυτή την πρόταση. Μάλιστα. Τώρα, μια κοινή τροπολογία που υπευλήθη από τα δύο σώματα της Γερμανικής Βουλής, από την Ρωμανική Βουλή, τη Ρωμανική Βουλή και το, την Κροτική Βουλή. Η κυρία Φλωρέα από την Ρουμανική Βουλή θα μας παρουσιάσει την πρόταση. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, εμείς είμαστε υπέρ της τροπολογίας 4, στο άρθρο 4, παράγραφος 2, που αφορά το δικαίωμα υποβολής ερωτήσεων. Θα θέλαμε να έχουμε μία προθεσμία έξι εβδομάδων για τις απαντήσεις που θα δίνει η Ευρωπόλ στις ερωτήσεις των μελών της μικτής ομάδας. Να υπάρχει προκαθορισμένο χρονικό πλαίσιο έξι εβδομάδων. Επίσης, το θέμα του παραδεκτού της ερώτησης να ελέγχεται από την τριάδα των προεδριών, την τρόικα προεδριών και όχι από τους συμπροέδρους της μικτής ομάδας. Καλύτερα τέσσερις να ελέγχουν το παραδεκτό και όχι μόνο δύο ή δύο συμπροέδροι. Νομίζω ότι έτσι ενισχύεται οι νομιμοποίηση των ερωτήσεων, της κρίσης του παραδεκτού μάλλον των ερωτήσεων. Επίσης θα θέλαμε οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις να αναρτώνται στο IPEX. γιατί με τον αυξανόμενο αριθμό των ερωτήσεων θα μπορούν έτσι τα μέλη να ενημερώνονται από το IPEX και να βλέπουν αν η ερώτηση έχει ήδη υποβληθεί, οπότε η απάντηση ήδη καλύπτεται. Η συγκεκριμένη τροπολογία τη χάνει της υποστήριξης και της γερμανικής και της κροατικής αντιπροσωπείας. Επίσης, Καλό θα ήταν οι ερωτήσεις αυτές να αποστέλλονται σε όλα τα μέλη της μικτής ομάδας, ώστε να τηρείται η αρχή της διαφάνειας. Η δεύτερη κοινή τροπολογία των τριών αντιπροσωπιών, γερμανικής, ρουμανικής και κροατικής, αφορά το σημείο 9, παράγραφος 5. Συγκεκριμένα, το διορισμό του εκπροσώπου στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπόλ. Με βάση την αρχή της αναλλαγής ε, της περιτροπής ε, της ε, Προεδρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και βάση της αρχής της ισότητας, της ισοτιμίας μεταξύ των κρατών μελών, θα θέλαμε όλα τα κράτη-μέλη να μπορούν στη διάρκεια της Προεδρίας να ορίσουν ένα μέλος που θα λαμβάνει μέρος στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπόλ για να μπορεί το κράτος μέλος να ενημερώνεται καλύτερα για τη συζήτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπόλ. Το άρθρο 5 είδαμε ότι τροποποιήθηκε και από άλλες αντιπροσωπείες με την ίδια ιδέα να διέπει τις τροπολογίες, δηλαδή την θητεία την πεντάμινη. Θα θέλαμε λοιπόν να ζητήσουμε από τις αντιπροσωπείες να υποστηρίξουν τη δική μας τροπολογία και να καταλήξουμε σε αιμοφωνία, σε συνένεση. Αν δεν καταστεί δυνατό κάτι τέτοιο, είμαστε ανοιχτοί και σε άλλες λύσεις. Όπως πρότεινε προηγουμένως και ο Διευθυντής του, Διοικη... του Διοικητικού Συμβουλίου. Γιατί το Προεδρείο του Διοικητικού Συμβουλίου απαρτίζεται από ένα τακτικό μέλος και ένα αναπληρωματικό μέλος από κάθε κράτος μέλος. Εμείς θα προτείναμε δύο μέλη, ένα τακτικό και ένα αναπληρωματικό και τους δύο συμπροέδρους, οπότε διασφαλίζεται η αρχή της συνέχειας. Γιατί έχουμε την πενταετή θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και τηρείται και η αρχή της διαφάνειας και οι υπόλοιπες αρχές που κατοχυρώνονται στον κανονισμό για την Ευρωπόλ. Αν και τα δύο μέλη, το τακτικό και το αναπληρωματικό, συμμετέχουν ε, στις συνεδριάσεις, τότε μόνο ένας θα δικαιούται να λαμβάνει το λόγο. Αλλά ανακύπτουν περιπτώσεις όπου οι, συ... οι συμπρόεδροι δεν μπορούν να είναι παρόντες και οι δύο ταυτόχρονα στις ε, συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Μάλιστα, Τώρα η Πορτογαλία, η Πορτογαλική αντιπροσωπεία. Κυρία Δίας Σίλβα θα μας παρουσιάσει την τροπολογία 6 της Πορτογαλίας. Ε. Ευχαριστώ, εδώ πέρα είμαι. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Θα μιλήσω πορτογαλικά μια και έχουμε διερμηνία για να σας παρουσιάσω την τροπολογία μου στο άρθρο 5 του κανονισμού. Αγαπητοί συνάδελφοι, όπως είπε πριν από λίγο η πρόεδρος, στην τελευταία συνεδρίαση στο Βουκουρέστι ε, καταλήξαμε σε ένα ακόμη αδιέξοδο σε ό,τι αφορά τον διορισμό του αντιπροσώπου του, της μικτής ομάδας στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπόλ. Τότε είχα προτείνει να μην ε, έχουμε το, το, κανόνα, το κανόνα της περιτροπής και γι' αυτό η Πορτογαλική Βουλή κατέθεσε μία πρόταση που ε, προσθέτει στο άρθρο 2 ε, του 5 ε, λέει ότι ο εκπρόσωπος της Ευρωπόλ στο Διοικητικό Συμβούλιο θα ορίζεται από αυτό που έχει την συμπροεδρία της μικτής ομάδας για μία εξάμηνη περίοδο και έτσι τηρείται η αρχή της εκπεριτροπής εκπροσώπησης. Θα θέλαμε να ληφθεί υπόψη αυτή η πρότασή μας, η τροπολογία, για να καταλήξουμε τελικά σε συμφωνία που κατά τη γνώμη μας είναι δίκαιη, ισορροπημένη και αφήνει ε, ικανοποιημένους τους πάντες χωρίς να περιθωριοποιεί κανένα. Σας ευχαριστώ. Thank you. And then House of ευχαριστώ. Μετά από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Κύπρου, ο κύριος Δημήτρης Δημητρίου, επικεφαλής της Αντιπροσωπείας. Ευχαριστώ. Η δική μας η τροπολογία για το άρθρο 5 στηρίζεται στην θέση αρχής που έχουμε εκφράσει και στο Βουκουρέστι τον Φεβρουάριο, αλλά και προηγουμένως όταν συζητήθηκε το θέμα. Και πιστεύουμε ότι ο εκπρόσωπος θα πρέπει να ορίζεται από το κράτος που προεδρεύει η χώρα του. Αν η χώρα αυτή πιστεύει στην ε, συνέχιση, το continuity και θέλει να ορίσει τον πρόεδρο, τον εκπρόσωπο, συγγνώμη, από την προηγούμενη χώρα και να διατηρήσει, έχει καλός. Ή αν θέλει, μπορεί να ορίσει ως εκπρόσωπο όποιο μέλος θέλει, ακόμη και μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Βασίζεται στη λογική ότι δίνει την ε, δυνατότητα στην χώρα που προεδρεύει να έχει τον πρώτο λόγο για το ποιο θα είναι ο εκπρόσωπος αυτός. Βλέπω ότι υπάρχει μια τάση για συνένεση ως προς αυτό και είμαι αισιόδοξο ότι σήμερα θα καταλήξουμε με ομοφωνία σε αυτό το ζήτημα. Ευχαριστώ. Thank ευχαριστώ. Από την Βουλή της Σουηδίας, ο κύριος Πέτερ Λέπερ επικεφαλής της Σουηδικής Αντιπροσωπεία. Τροπολογίε 11 και 13. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Όσον αφορά τι διατάξεις περί διορισμού στο ΔΣ της Europol, το άρθρο 5 λέει πως θα υπάρξει μία αυτόματη διαταγή για τον διορισμό στο ΔΣ του της Γεροπολ. Δεν χρειαζόμαστε κάθε φορά συνεδρίαση, ανταυτού μπορεί να αφιερώνει το χρόνο στην κύρια δουλειά μας. Θα πρέπει η σειρά αυτή να σχετίζεται με την εναλλασσόμενη Προεδρία, έτσι ώστε να αποτελεί ε, ακριβώ ο παρατηρητής αυτός κάθε ε, των καθηκόντων της. Κατά την απόψή μας λοιπόν είναι σημαντικότερο όλα τα εθνικά κοινοβούλια και αντιπροσωπείες να έχουν ίση ευκαιρία να σχηματίσουν ίδιαν άποψη για το τι περιλαμβάνει αυτή η δουλειά και να έχουν μια εικόνα για το πώς λειτουργεί όντως το ΔΣ της Europol. Βεβαίω το όφελος αυτό της αυτόματης ε, διαδοχής ε, θα έλυνε και το ζήτημα της λήψης αποφάσεων. Θα ήθελα να πω επίσης ε, λίγα λόγια για ένα άλλο ζήτημα το οποίο μας απασχολεί αφορά τις διατάξεις περί θέσεως ενισχύ και αναθεώρησης του κανονισμού. Προτείνουμε να αλλάξουν να αλλάξει το άρθρο 6 εδάφιο 1 έτσι ώστε οι σχετικές αλλαγές να τίθενται ενισχύει λίγο καιρό αργότερα. Έτσι ώστε μια τροπολογία η οποία εγκρίνεται κατά τη διάρκεια της ε, συνεδρίασης να αφορά ένα θέμα το οποίο ε, συζητιέται στην ίδια συνεδρίαση. Τέλος, προτείνουμε αναθεώρηση του άρθρου 6 εδάφιο 2 που αφορά την ε, διαδικασία για την αναθεώρηση του κανονισμού και την εξέταση των προτάσεων. Η ομάδα αυτή της εξέταση είναι ακόμη στις πρώτες μέρες της και είναι λογικό να χρειαστεί να δούμε διάφορες ε, διαδικασίες και το αποτέλεσμα αυτής ε, της διαδικασίας δεν είναι ακόμα γνωστό, οπότε θα πρέπει ακριβώς να έχουμε μια τέτοια προσέγγιση προς τον κανονισμό. Καλό είναι να διατηρηθούν οι διαδικασίες οι οποίες λειτουργούν αποτελεσματικά, ενώ οι υπόλοιπε να διαγραφούν. Σα Σας ευχαριστώ και τώρα η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα μας την παρουσιάσει ο κ. Πίτερ, που είναι αντιπρόεδρος της αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Μικτή Ομάδα. Τροπολογία 12. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα σας παρουσιάσω τη θέση της αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Μικτή Ομάδα σε ό,τι αφορά το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπόλ. Η θέση μας είναι ξεκάθαρη η επιλογή του εκπροσώπου θα πρέπει να γίνεται μεταξύ των τακτικών μελών, συμπεριλαμβανομένων του εκπροσώπου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, για 18 μήνε με μία παράταση άλλο ένα Ε, για το άρθρο 3.2, η τροπολογία της Ολλανδίας ε, δεν μας βρίσκει σύμφωνος. Διαφωνούμε με την Ολλανδική τροπολογία. Σε ό,τι αφορά την ε, τροπολογία 2, για το 4.1α, Εκεί συμφωνούμε εν μέρη με τη σχετική τροπολογία και έχουμε και κάποιες ερωτήσεις για το τι νόημα ακριβώ έχει το σημείο που λέει ότι η νέα έννοια επερωτήσεις διαδικαστικού χαρακτήρα. Αυτό το νέο στοιχείο μας προβληματίζει. Δεν ξέρουμε τι ακριβώς εννοεί. Θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε, αλλά αυτή η ιδέα των διαδικαστικών ερωτήσεων μα προβληματίζει και θα θέλαμε εξηγήσει. Σε ό,τι αφορά την τροπολογία 3 για το άρθρο 4.1.ε, εκεί η αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διαφωνεί ριζικά με τη σχετική τροπολογία. Και μάλιστα έγινε σχετική συζήτηση τον Απρίλιο του 2017 στην Πρατισλάβα και δεν μπορούμε να δεχτούμε την τροπολογία αυτή. Σε ό,τι αφορά την τροπολογία 4 για το άρθρο 4.2 το δικαίωμα υποβολή ερωτήσεων. Η αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα μπορούσε να δεχτεί καταρχήν ένα τμήμα τη τροπολογίας, αλλά ίσως δεν χρειάζεται να αλλάξουμε τον εσωτερικό κανονισμό, γιατί υπάρχει μια σχετική κατευθυντήρια γραμμή που ε, εστάλει την περασμένη εβδομάδα στα κράτη-μέλη και πολλά στοιχεία αυτής της κατευθυντήριας γραμμής ε, ε, καλύπτουν την τροπολογία. Οπότε ίσως δεν χρειάζεται να τροποποιηθούν στο σημείο αυτό οι κανόνες του εσωτερικού κανονισμού. Επίσης, άρθρο 4.2, ε, ε, τροπολογία 5. Είμαστε υπέρ κάποιων τμήματων της τροπολογίας καταρχήν, αλλά το κείμενο γενικώ δεν μας βρίσκει σύμφωνος και για την τροπολογία 13, την τροπολογία για το άρθρο 6, τελικές διατάξεις, εκεί η αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διαφωνεί με την τροπολογία 13 της Σουηδίας. Και αυτή είναι η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη Μικτή Ομάδα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Έχουμε και πολλές γραπτές προτάσεις για την αλλαγή του εσωτερικού κανονισμού. Θα ακούσουμε ενδεχομένω αντιπροσωπείς που θέλουν το λόγο και για τα θέματα αυτά. Δύο λεπτά το πολύ για την κάθε αντιπροσωπεία. 8 λεπτά συνολικά. Τέσσερις είναι αντιπροσωπείε. Θα σα δώσω το λόγο με τη σειρά που υποβάλλατε και τις γραπτές σα προτάσεις. Πρώτα θα δώσω το λόγο στην Ουγγρική Αντιπροσωπεία, τον κύριο Ιστον Κεντάνη. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. ε, ως επικεφαλής αντιπροσωπής της Ουγγαρίας στη μεικτή ομάδα και σε σχέση με την ε, επιστολή της 17ης Μαΐου για το διορισμό του εκπροσώπου της Μικτής ομάδας στην ε, συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπόλ. Σας ευχαριστώ καταρχήν που ε, συγκαλέσατε αυτή τη συνεδρίαση και λάβατε υπόψη στο έτοιμά μας όπως και η βουλγαρική και η ρωμανική αντιπροσωπεία, θα θέλαμε ε, η διάρκεια της εντολής ε, να είναι αντικείμενο συνένεσης πιο μακροχρόνιας. Και θα μπορούσαμε να δεχτούμε το διορισμό αρκεί να τηρείται η αρχή της συνέχειας και της διάρκειας γιατί έχουμε την τριάδα των προεδριών που καλύπτουν μια περίοδο 18 μηνών, οπότε καλό ήταν να ευθυγραμμιστούμε με αυτό το 18 μηνό και για την ε, εντολή του εκπροσώπου. Ευχαριστώ. Μετά ο κύριος Μύρουσλαβ είναι από την Τσεχική Γερουσία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να συμφωνήσω με τον κύριο Μπζόχ ε, από την Τσεχική Βουλή. Συμφωνούμε σε όλα, εκτός ε, από το ότι η μεικτή συνέλευση προσωπείται από τον αντιπρόσωπο της προεδρεύουσας χώρας ή από ένα μέλος ε, της Τρόικας για 18 μήνες. Εμείς προτείνουμε 12 μήνες και επίσης στηρίζουμε την αλλαγή του κανονισμού που θα μας φέρει πιο κοντά στον μηχανισμό COSAC και ελπίζουμε να μπορέσουμε να βρούμε κάποια συνένεση. και να μην χρειάζεται να ψηφίζουμε πολύ συχνά. Σας ευχαριστώ και μετά από την Ιρλανδία Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας ε, συμβουλεύσω για το θέμα της επιλογής ε, των μελών της Μεκτής ε, Συνέλευσης στο θέμα ακριβώς ε, τη αντιπροσώπευση τη Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων τη ε, Ιρλανδίας. Ε, η άποψή μας είναι πως οι εκπρόσωποι στο Διοικητικό Συμβούλιο θα πρέπει να ορίζονται από την κοινοβουλευτική αντιπροσωπεία του κράτους μέλους που έχει την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα η εντολή θα πρέπει να περιορίζεται στην εξάμεινη θητεία της Προεδρίας με την δυνατότητα παράτασης ε, υπό ορισμένες συνθήκες εάν παραδείγματο χάρη μια χώρα ε, που θα έχει την Προεδρία θέλει, δεν θέλει να αναλάβει αυτήν την θέση. Θεωρούμε ότι είναι η πιο δίκαιη λύση καθώς δίνει σε κάθε κράτος μέλος την ίδια δυνατότητα συμμετοχής ε, στο ΔΣ και η πιο διαφανής ε, προσέγγιση και θα δώσει τη δυνατότητα στι εθνικέ αντιπροσωπείε να προγραμματίζουν και να ξέρουν πότε θα αναλάβουν τον ρόλο αυτόν. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Μετά έχουμε τις γραπτές παρεμβάσεις από την ε, Σλοβενία. Δεν υπάρχει κάποια παρουσίαση. Είναι εδώ. Τώρα συνεχίζουμε με την ανταλλαγή απόψεων στις προτινόμενες αλλαγές του κανονισμού. Έχουμε πολλούς ομιλητές που θέλουν το λόγο. Ο κύριος Απέλ από την Πολωνία. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ. Είναι σημαντικό να έχουμε μια αποτελεσματική και διαφανή διαδικασία. Γι' αυτό η Πολωνία είναι υπέρ της άμεσης απάντησης των ερωτήσεων από την Ευρωπόλ, όσο γίνεται πιο γρήγορα. Αλλά θέλουμε να είναι και αποτελεσματική η Ευρωπόλ ώστε ε, και ο αποσπασμένος αξιωματούχος να έχει το χρόνο να εγκληματιστεί στην Ευρωπόλ. Σίγουρα αυτά ακούγονται απλά, αλλά δεν είναι καθόλου απλά. απλά. Γι' αυτό είμαστε υπέρ της 18μηνης ε, εντολής για την άσκηση της ε, θητείας του εκπροσώπου της μικτής ομάδας. Thank Σε ευχαριστώ. Και μετά ο κύριος Ήρμερ από την Γερμανία. Ναι, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πολύ. Εμείς αναφερόμαστε στο 4.1 του ιστορικού κανονισμού. Θα θέλαμε τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, δηλαδή εμείς, να συμμετέχουμε στο ε, σχέδιο ημερήσιας διάταξης, να κάνουμε προτάσεις, να μπορούμε να υποβάλουμε προτάσεις, ειδικότερα όσον αφορά την αποδοχή ή τη διαγραφή σημείων στην ημερήσια διάταξη μέχρι δύο εβδομάδες πριν τη συνεδρίαση. Επιπλέον, θα θέλαμε να υπάρχει δυνατότητα να μπορούμε να αλλάξουμε την ημερήσια διάταξη σε διάρκεια συζήτηση. Όπω για παράδειγμα, αν στο τέλο μια συνεδρίαση κάποιο σημείο προκύπτει ω σημαντικό, αλλά λόγω προθεσμιών δεν έχει συμπεριληφθεί, να μπορούμε να υποβάλουμε ένα αίτημα να ε, εξεταστεί νωρίτερα. Γι' αυτό λοιπόν θα είχε νόημα να μπορούμε να αλλάξουμε έτσι και να ψηφίσουμε ε, την αλλαγή μια ημερησία διαταξία. Θέλαμε δηλαδή ω μέλη τη Επιτροπή Ελέγχου να έχουμε περισσότερε δυνατότητε να παρέμβουμε στην ημερησία διαταξιά. Αυτή είναι η πρότασή μα όσον αφορά την αλλαγή του άρθρου 4.1. Thank you. And then Daly. Ευχαριστώ κυρία Νταλή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η κυρία Ντέιλι. Ο κύριος Λάνετ από την Εστονία. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Όσον αφορά τον ε, διορισμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και την διάρκεια της αιτίας τους. Κατά προτίμηση θα έπρεπε να είναι ένας πρόσωπος ε, της ε, Τρόικας, της Προεδρίας και να διορίζεται για 18 μήνες. Γιατί? Γιατί άπαξ και οριστεί από την Επιτροπή μας το άτομο αυτό θα πρέπει να μάθει πώς λειτουργεί το ΔΣ και να μπορέσει να συνεισφέρει και αποτελεσματικά. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Χαρακόπουλος από την Ελλάδα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η συμμετοχή εκπροσώπου της ΜΟΚΕ ως παρατηρητής της συνεδριάσης του Διοικητικού Συμβουλίου της Europol είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για την ενημέρωσή μας. Λόγω του εξειδικευμένου χαρακτήρα του αντικειμένου και προκειμένου ο εκπρόσωπος της ΜΟΚΕ στο Διοικητικό Συμβούλιο της Europol να αποκτήσει μεγαλύτερη εμπειρία και καλύτερη γνώση του αντικειμένου επιβάλλεται να βρεθεί η χρυσή τομή για τη διάρκεια της θητείας του. Ως επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας πιστεύω ότι η 12μηνη θητεία είναι ισορροπημένη χρονικά καθώς ο εκπρόσωπος θα έχει αποκτήσει εμπεριστατωμένη άποψη και γνώση του αντικειμένου αφετέρου θα παράσχει στη ΜΟΚΕ τη σχετική πληροφόρηση για τα θέματα αρμοδιότητας του Διοικητικού Συμβουλίου. Το δεύτερο στο οποίο θα ήθελα να αναφερθώ είναι ο τρόπος λήψεως των αποφάσεων με συνένεση ομοφωνία, όπως προβλέπεται στον κανονισμό λειτουργίας. Αναμφίβολα η συνένεση αποτελεί βασική αρχή της συνεργασίας και κατά συνέπεια θα πρέπει να διαφυλαχθεί. Ακόμη και όταν υπάρχουν διαφωνίες, όπως συνέβη στην τελευταία συνεδρίαση της ΜΟΚΕ στο Βουκουρέστι για τη διάρκεια της θητείας του εκπροσώπου, ο στόχος μας θα πρέπει να είναι η επίτευξη ομοφωνίας μέσα από τη διαδικασία της συζήτησης και τον συγκερασμό των απόψεων. Σε περίπτωση όμως αδυναμίας επίτευξης πλήρους ομοφωνίας υπάρχει, όπως ελέγχθη, δυνατότητα προσφυγής σε ψηφοφορία και λήψη αποφάσεων με ενισχυμένη πλειοψηφία τριών τετάρτων επί των ψηφισάντων, όπως προβλέπεται και στην ΚΟΖΑΚ. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και τέλος ο κύριος Σαμπατόσκος από τη Λιθουανία. sorry. Lietuvos delegacija siūlo palaikyti vis tik tai 18 mėnesių. Ευχαριστώ πολύ. Η λιθανική αντιπροσωπεία θα ήθελε να υποστηρίξει το την περίοδο των 18 μηνών. για εκπροσώπους στο Διοικητικό Συμβούλιο διότι η συμμετοχή της Τριάδας Προεδριών είναι πολύ σημαντική στο Διοικητικό Συμβούλιο. Θα μας βοηθήσει να διασφαλίσετε η συνέχεια. Δεν καταλαβαίνουμε ακριβώς την πρόταση των 12 μηνών σε τέτοια περίπτωση το ερώτημα είναι ποιος θα εκπροσωπείται. Η σημερινή Προεδρία, η τρέχουσα Προεδρία, η παρελθούσα ή η μελλοντική Προεδρία. Η προηγούμενη δηλαδή ή η επόμενη ή η τρέχουσα. Και η περίοδος των 12 μηνών κατά την άποψή μας δεν είναι αρκετά μεγάλη. Θα είναι αδύνατο να διασφαλιστεί η συνέχεια. Οπότε προτείνουμε εμείς 18 μήνες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ αγαπητά μέλη, ευχαριστώ πολύ για τις τροπολογίες σας, τις συμμετοχές σας και τα σχόλιά σας. Θα συνεχίσουμε τη συζήτησή μας αύριο. Τώρα πάμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης ανταλλαγή απόψεων με τον κύριο Βιβιορόφσκι, Ευρωπαίο ε, επόπτη προστασία δεδομένων και τον καθηγητή Φρανσο Πελεγκρίνη, πρόεδρο του ε, Συμβουλίου Συνεργασίας της Ευρωπόλου. So please, Παρακαλώ, έχουμε φτάσει στο τελευταίο μέρος της απογευματινής μας ε, συνεδρίασης ε, πριν από την εκδήλωση που θα ξεκινήσει στις 7 στο νίκο της Ευρωπαϊκής Ιστορίας. Αλλά πριν από αυτό έχουμε ένα σημείο επί της ουσίας. Αφορά την αναφορά από τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων και το Συμβούλιο Συνεργασίας ε, της Ευρωπόλ. Δύο σημαντικά ζητήματα. Έχουμε εδώ δύο μιλητέ ε, που ε, βρίσκονται ήδη εδώ στο βήμα. Ο βοηθός Επόπτη Προστασίας Δεδομένων, ο κύριος Βιβγερόφκη και ο κύριος Πελεγκρίνη. Αλλά πριν παρουσιάσουν αυτά που έχουν να μας πούν και παρακαλώ να έχω την προσοχή σας, θα ήθελα να κάνω κάτι το οποίο αναγκάστηκα να κάνω δυστυχώς ως πρόεδρος της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ της ε, Επιτροπής ε, αυτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην πρώτη ευκαιρία που είχαμε στην πρώτη τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ μετά τις θερινές διακοπές που είναι τώρα διότι στις θερινές διακοπές είχαμε δυστυχώς ε, μια πολύ άσκημη είδηση για τον θάνατο του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων την τελευταία πενταετία του κυρίου Τζάνι Μπουταρέλη. Ήταν πρώτο βοηθός ε, επόπτη προστασίας δεδομένων του Πίτερ Χάστινγκς υπό την ιδιότητά του ως βοηθός και μετά ως επόπτης, Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων. Ο ίδιος ερχόταν τακτικά στις συνεδριάσεις ε, της ε, Επιτροπής ΛΥΜΠΕ αντίλασε ε, συχνά απόψεις με μεγάλη ένταση για πολλά χρόνια με την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ και στάθηκε στο ως ένα εκπρόσωπος φορέα που ασχολείται με την προστασία, το απόρριτο και την ασφάλεια των Ευρωπαίων πολιτών ενώπιον των ευρωπαϊκών θεσμών, συμπεριλαμβανομένου του Κοινοβουλίου μα, προστατεύοντα έτσι τα θεμελιώδη δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών όπω θεσπίζονται στο χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό το λόγο, πριν ξεκινήσουμε με αυτήν εδώ, αυτό εδώ το κομμάτι τη συνεδρίαση, ζήτησα ενό λεπτού σιγή για να αποτίσουμε φόρο τιμή στον Τζάνι Μπουταρέλη, ο οποίο επιτέλεσε τα καθήκοντά του μέχρι την τελευταία στιγμή της ζωής του. επιτέλεσε επάξια χάρη στην ε, προσωπική του ικανότητα να φέρνει αποτελέσματα ακόμη και όταν ε, δυστυχώς ε, έφτανε στο τέλος της ζωής του με τόσο λυπηρό τρόπο. Αποτίσαμε φόρο τιμή στη μνημή του σε μια διάσκεψη που έλεγε χώρα στις Βρυξέλλες και θα πρότεινα να αποτίσουμε τιμή στη μνήμη του με ενός λεπτού συγγύη πριν ξεκινήσουμε αυτό το σημείο της ημερησίας διάταξης. Σα Σας ευχαριστώ πολύ για αυτό το λεπτό που αφιερώσαμε για να εκφράσουμε το σεβασμό μας. Και προχωράμε στο επόμενο σημείο λοιπόν, σε αυτό το σημείο τη ημερήσιας διάταξης ε, είναι αυτό στο οποίο θα έχουμε δύο παρουσιάσει από τα μέλη του πάνελ εδώ από τον βοηθό Ευρωπαίο Επόπτη Προστασία δεδομένων τον κύριο Βιβερόφσκι και από τον καθηγητή κύριο Πελεγκρίνη. Θα ήθελα να σας θυμίσω ότι ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων είναι το θεσμικό όργανο που παρακολουθεί και διασφαλίζει την υλοποίηση του κανονισμού Ευρωπόλ σε σχέση με την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων των Ευρωπαίων πολιτών, ειδικότερα εκείνων που ε, τους οποίους αφορά η επεξεργασία δεδομένων και το ε, Συμβούλιο Συνεργασίας της Ευρωπόλ είναι το συμβουλευτικό όργανο για αυτό το θέμα. Συγκεντρώνει τις Εθνικές Εποπτικές Αρχές, τον EDPS, εκδίδει γνωμοδοτήσεις και συστάσεις. Η συνεργασία μεταξύ Ευρωπόλ και Ευρωπαϊκού Επόπτη Προστασίας Δεδομένων και Συμβουλίου Συνεργασίας μέχρι στιγμής ε, ε, λειτουργεί ομαλά, όπως ακούσαμε στην τελευταία συνεδρία στο Φεβρουάριο ε, του EDPS. Αυτό το εκτιμάμε ιδιαίτερα δεδομένη τη σπουδαιότητα τη επεξεργασία δεδομένων. Αλλά α ακούσουμε τι εκθέσει που αφορούν το τελευταίο εξάμεινο συνεργασία. Θα ακούσουμε πρώτα απ' όλα λοιπόν τον κύριο Βιβιερόφσκι, τον οποίο θα ακολουθήσει ο κύριος Πελεγκρινή και ανακοινώνω ότι θα έχουμε ένα γύρο έρωτα απαντήσεων Προτείνω λοιπόν να, αν θέλετε να μιλήσετε, να το δηλώσετε εγγράφως σε αυτά τα χαρτιά, σε αυτά τα έγγραφα και θα μιλήσετε αμέσως μετά τις δύο παρουσιάσεις. Κύριε Βιβιερόσκη, σας προτείνω να ε, πάρετε 12 λεπτά για την παρουσίασή σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε και κυρία Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη των Εθνικών Κοινοβουλίων και μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είναι τιμή μου και προνόμιον που βρίσκομαι εδώ για να σας αναφέρω τις δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Επόπτη Προστασίας Δεδομένων για τους τελευταίους μήνες μετά από την τελευταία μας συνεδρίαση. Παρότι φυσικά θα προτιμούσα να μην έπρεπε να το κάνω εγώ να ήταν εδώ ο Τζοβάνι Μπουταρέλη όπως έκανε συνήθως ε, στις ε, συνεδριάσεις της ομάδας. Βλέπω πολλούς από τους ανθρώπους που λάμβαναν μέρος στις συναντήσεις της ομάδας, αλλά και νέα μέλη του Ευρωκοινοβουλίου. Θα ήθελα λοιπόν να τονίσω για άλλη μια φορά ότι ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων ασχολείται με την προστασία δεδομένων και τα σχετικά ζητήματα που σχετίζονται με όλα τα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δυνάμει του κανονισμού συνήθως που εκδίδεται για τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και που μοιάζει με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων. Αλλά σε αυτή την περίπτωση υπάρχει ένα ειδικό μέρος των κανόνων που προέρχεται από τον κανονισμό της Ευρωπόλ. Ταυτόχρονα αυτό γίνεται σε συνεργασία με τις Εθνικές Αρχές Προστασίας Δεδομένων για προφανείς λόγους. Ε, ποπτεύουμε τον ίδιο τον οργανισμό, ενώ τα περισσότερα δεδομένα που έχει στα χέρια του οργανισμού Αυτό προέρχονται από τι εθνικέ αρχέ και διαβιβάζονται, ε, συγγνώμη, πρώτα απ' όλα δημιουργούνται και ε, υφίστανται επεξεργασία σε εθνικό επίπεδο και πολλές φορές τα αποτελέσματα αυτών καταλήγουν στο επίπεδο ε, της Ευρωπόλ. Οπότε υπάρχει εποπτεία σε όλα αυτά τα επίπεδα και από την 1η Μαΐου του 2017 προσπαθούμε να κάνουμε όλη αυτή την εποπτεία μαζί σε όλα τα επίπεδα. Ευχαριστούμε για το φόρο τιμής στον Τζοβάνι Πουταρέλη και ήθελα να σας διασφαλίσω ότι θα υπάρξει συνέχεια της δουλειάς ε, του EDPS ε, όπως είχε προβλεφθεί στον κανονισμό για τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ εξελέγγυρ μαζί με τον Τζοβάνι Μπουταρέλη για την ίδια θητεία μέχρι τις 5 Δεκεμβρίου φέτος. Και μέχρι τις 5 Δεκεμβρίου του 2019 το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο θα πρέπει να εκλέξουν νέο Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων. Οι δυσκολίες ε, τη εποπτεία ε, και σε επεξεργασία των δεδομένων στον τομέα τη επιβολή του νόμου σα είναι γνωστέ. Δεν θα σπαταλήσω το χρόνο σα για να τι ξανατονίσω. Απλά θα ήθελα να τονίσω το γεγονό ότι η βάση δεδομένων και η πόροι είναι όλο και μεγαλύτερη ε, στα χέρια των αρχών της επιβολής του νόμου και τα συστήματα πληροφορικής που χρησιμοποιούνται ε, τείνουν να γίνονται όλο και πιο περίπλοκα. Φυσικά τα συστήματα πληροφορικής ε, που χρησιμοποιούνται από την Ευρωπόλ χρησιμεύουν ταυτόχρονα στην Ευρωπόλ και στους στόχους της, αλλά και στην συνεργασία των αστυνομικών αρχών και των αρχών επιβολής του νόμου στις επιμέρους χώρες. Οπότε ε, είναι δύο πλευρές του ίδιου νομίσματος. Η συνεργασία με το Συμβούλιο Συντονισμού που θα σας παρουσιάσει ο κύριος Πελεγκρίνη Μα δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε αυτό την εποπτεία σε όλα τα επίπεδα. Οι δραστηριότητες των τελευταίων λίγων μηνών, οι πιο σημαντικές, μπορούν να χωριστούν σε δύο κατηγορίες. Έχουμε το κομμάτι της συνεργασία και τις εποπτικές ε, ε, δραστηριότητες. Το κομμάτι της συνεργασίας συνίσταται στην σχεδόν καθημερινή συνεργασία με την Ευρωπόλ και τις ομάδες εκεί τις ομάδες που ασχολούνται με την προστασία των δεδομένων απευθείας και εκείνων που ασχολούνται με τα συστήματα πληροφορικής ε, που χρησιμοποιεί η Ευρωπόλ. Η βασική δομή εδώ βασίζεται σε μηνιαίε συναντήσει που οργανώνονται από τον EDPS ε, ή την Ευρωπόλ. Στις συνεδρίες αυτές προσπαθούμε να προβλέπουμε και τι πρέπει να θυμόμαστε για τις εβδομάδες που ακολουθούν. Οι εποπτικές αρχές, ωστόσο, είναι πιο χρονοβόρες για μας. Ξεκινούν με τις πληροφορίες που πρέπει να ε, παρέχει η Ευρωπόλ στις εποπτικές αρχές που προέρχονται από τις επιχειρησιακές δραστηριότητες, ε, πιθανές παραβιάσεις δεδομένων και πιθανές ε, διαβιβάσεις σε τρίτες χώρες. Τα έργα επιχειρησιακής ανάλυσης είναι τα κύρια κομμάτια της δραστηριότητας της Ευρωπόλ που μας απασχολούν. Καθένα από αυτά τα έργα επιχειρησιακής ανάλυσης ε, ε, εστιάζεται σε συγκεκριμένο τομέα εγκληματών όπως παιδική πορτογραφία, οργανωμένες εγκληματικές ομάδες, ε, τρομοκρατία και η Ευρωπόλ πρέπει να ενημερώνει τον EDPS κάθε φορά που ανοίγει, τροποποιεί ή κλείνει κάποια επιχειρησιακή δραστηριότητα. Σε περίπτωση παραβίαση δεδομένων, οι πληροφορίε αυτέ πρέπει να παρέχονται σε σχέση με ένα τέτοιο γεγονό στον EDPS. όπω ε, αναφέρεται στον κανονισμό, εν χρόνο. Δεν υπάρχει χρονικό όριο όπω υπάρχει στο GDPR για αυτό, αλλά εμεί λαμβάνουμε τι πληροφορίε αυτέ χωρί καθυστέρηση από την Ευρωπόλη η μεταβάση δεδομένων σε τρίτες χώρες που ούτε είναι κατάλληλες ούτε έχουν επιχειρησιακή συμφωνία για ανταλλαγή δεδομένων σε εξαιρετικέ περιπτώσει, όπω για παράδειγμα για την υποστήριξη ορισμένων ερευνών, διαβίβαση δεδομένων εκτό τη Ευρωπόλ. Αυτό ε, πρέπει να ακολουθείτε, να συνοδεύεται από ενημέρωση του EDPS έχουμε τις γενικές διαβουλεύσεις όπου καταστάσεις προσπαθούμε να βοηθήσουμε την Ευρωπόλ στις γενικές δραστηριότητες του θεσμού. Οι διαβουλεύσεις, παραδείγματα τέτοιων διαβουλεύσεων από τον περασμένο μήνα, από τους περασμένους μήνες είναι ε, οι διευθετήσεις ε, συνεργασίας με τρίτες χώρες ε, όπου καθορίζονται οι προϋποθέσεις ανταλλαγής προσωπικών δεδομένων ε, και πώς αυτό γίνεται σε περίπτωση που η Ευρωπόλ χρειαστεί να χρησιμοποιήσει μια από τις εξαιρέσεις που προβλέπονται στον κανονισμό Ευρωπόλ υπό το άρθρο 25. Τώρα από τον Μάρτιο του 2019 προσπαθούμε να αξιολογούμε όλα τα πιθανά σενάρια που σχετίζονται με τον Brexit συμπεριλαμβανομένου ειδικότερα του πολύ δυστυχούς ενδεχόμενου να έχουμε ένα Brexit χωρίς συμφωνία, no deal Brexit όπως ονομάζεται, που θα δημιουργήσει διάφορα προβλήματα πρόσβασης δεδομένων στην Ευρωπόλ και για τις αρχές του νόμου Βασιλείου. Εμείς προσπαθούμε να προετοιμάσουμε λύσεις που ενδεχομένως θα μπορούν να λειτουργήσουν από την πρώτη ημέρα και αφορούν τη μελλοντική συνεργασία των ε, οργανισμών αυτών, των οντοτήτων αυτών. Οι κανόνε φυσικά αυτή τη συνεργασία ε, συντάσσονται από την Ευρωπόλη και το Διοικητικό του Συμβούλιο, αλλά προσπαθούμε να βοηθήσουμε και εμεί αυτό το κλάδο. Ένα άλλο παράδειγμα υποδιαβούλευση ε, με τις εποπτικέ αρχές είναι το πρόβλημα των ε, μονάδων οικονομικών πληροφοριών. Προσπαθούν να βρουν του αλληλοσχετισμού μεταξύ ύποπτων οικονομικών συναλλαγών και υποκείμενων εγκληματικών δραστηριοτήτων, ούτω ώστε να προλαμβάνουν και να καταπολεμούν το ξέπλυμα μαύρου χρήματο. Η ανταλλαγή πληροφοριών είναι οργανωμένη σε όλα τα επίπεδα. Μέσω του ViewNet και με την Ευρωπόλ και συζητάμε τη μελλοντική λύση, τη μελλοντική πρόταση που θα έχουμε τόσο με τον ίδιο το θεσμό όσο και με τις εποπτικές αρχές της χώρας. Επειδή διαπιστώσαμε ότι υπάρχουν μεγάλες διαφορές όσον αφορά τον ορισμό ενός υπόπτου, διότι μόνο οι ύποπτοι, αυτοί που έχουν οριστεί ως ύποπτοι μπορούν να αποτελέσει το αντικείμενο επεξεργασία δεδομένων με αυτόν τον τρόπο. Νομίζω θα το αναφέρει και ο κ. Πελεγκρίνη. Επίση, έχουμε και διαβουλεύσει κάθε φορά που Ευρωπόλ θα έχει μια νέα διαδικασία επεξεργασία δεδομένων με, δυνατότητα σημαντικού, με πιθανότητα σημαντικού κινδύνου. Εκεί πρέπει να γίνεται εκτίμηση κινδύνου για τα δεδομένα και τέτοιες περιπτώσεις, τέτοιες, ε, τέτοια σενάρια θα πρέπει να ε, σε τέτοια σενάρια θα πρέπει να γίνονται διαβουλεύσει. Είχαμε πέντε τέτοιε διαβουλεύσει με τον EDPS πέρυσι. Η τελευταία γνωμοδότηση ήταν το Σεπτέμβριο φέτο αφορούσε τι προποθέσει πρόσβαση τη Ευρώπολ στα προσωπικά δεδομένα επιβατών σύμφωνα με τη σχετική οδηγία. PNR όπω ονομάζεται. επίση ξεκινάμε έρευνε βάσει δική μα πρωτοβουλία για ζητήματα τα οποία έρχονται σε δική μα γνώση κατά τη διάρκεια των εποπτικών μα δραστηριοτήτων. Το 2019 έχουμε ξεκινήσει ήδη τέσσερις έρευνες τέτοιου είδους. Καταγγελίες. Πρέπει να παραδεχτώ ότι μου κάνει έκπληξη το χαμηλό ποσοστό καταγγελιών που έρχονται στον EDPS. Μέχρι στιγμής έχουμε λάβει μόνο δύο ε, παραδεκτές ε, καταγγελίες, ε, οι οποίες βρίσκονται υπό διερεύνηση στα γραφεία μας. Και τέλος, επιθεωρήσεις είναι το τελευταίο κομμάτι της παρουσίασής μου σήμερα. Φυσικά ο ακρογωνίος λήθος της δραστηριότητας του EDPS όσον αφορά την εποπτεία είναι η επιθεωρήση. Εμείς πραγματοποιούμε επιθεώρηση των νομικών ε, πτυχών της επεξεργασίας δεδομένων. Μέχρι στιγμής έχουμε κάνει τρεις ετήσιες επιθεωρήσεις και η τελευταία που έγινε τον Ιούνιο υπέστη επεξεργασία ε, τα έγγραφα υπέστησαν επεξεργασία στο γραφείο του EDPS με εστίαση στην επεξεργασία δεδομένα, δεδομένων στη χρηματοδότηση τρομοκρατίας, ε, χρηματοδότηση ε, ξέπνο μαύρου χρήματος, παράνομες ε, δραστηριότητες στο Darknet, ε, διαβίβαση δεδομένων σε τρίτες χώρες και νέες πρακτικές των κράτων μελών αποστολής μεγάλων ποσοτών δεδομένων στην Ευρωπόλ και τα αποτελέσματα με τα όλο και περισσότερα προσωπικά δεδομένα που έχουν στη διάθεσή τους οι εθνικές ε, αστυνομικές αρχές σε εθνικό επίπεδο στο πλαίσιο ποινικών ερευνών. Επίσης, ε, ε, βλέπουμε τις μεθοδολογίες που χρησιμοποιεί η Ευρωπόλ και τις παλιότερες συστάσεις μαζί με τους εμπειρογνώμονες από τις Εθνικές Αρχές Προστασίας Δεδομένων που καλούνται να συμμετέχουν. Η επιθεώρηση ελέγχου έχει εισταλεί στον εκτελεστικό διευθυντή της Ευρωπόλ, στην εκτελεστική διευθύντρια της Ευρωπόλ και κοινοποιήθηκε και στο Συμβούλιο Συντονισμού. Επίσης έχουμε μια μεγάλη στοχευμένη επιθεώρηση που θα σας ενδιαφέρει. Είναι η στοχευμένη επιθεώρηση του ε, προγράμματος TFTP που προσπαθεί να βρει ε, τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Μια συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, η χνηλάτηση της χρηματοδότησης της ε, τρομοκρατίας με αντικείμενο την επαλήθευση του ρόλου που έχει η Ευρωπόλη υπό τη συμφωνία στη FTP αφορά την επαλήθευση των ε, ετοιμάτων που αποστέλλονται στο προνομαζόμενο SWIFT. Η Ευρωπόλη δεν έχει πρόσβαση στη, σε επικοινωνία αλλά στα αιτήματα που αποστέλλονται. Έχουμε στείλει 8 ε, συστάσεις για περαιτέρω βελτίωση της επαλήθευσης των στοιχείων που χρησιμοποιούνται στην Ευρωπόλ. Η έκθεση αρχικά ήταν ε, απόρριτη ως EU Secret λόγω των προσδοκιών της αμερικανικής πλευράς. Αλλά μόλις ε, έχει πραγματοποιηθεί άρση του απορρίτου και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του DPS μέσα στις επόμενες ημέρες, μαζί με τις συστάσεις, με την εξαίρεση μίας σύστασης που εμείς αποφασίσαμε να παραμείνει απόρριτη λόγω του τεχνικού της ε, χαρακτήρα. Ο EDPS θα παρακολουθεί στενά την υλοποίηση αυτών των συστάσεων κατά τη διάρκεια των επιθεωρήσεων αυτών. Αυτά είναι τα σημαντικότερα από όσα συνέβησαν τους τελευταίους μήνες. Είμαι έτοιμος φυσικά να απαντήσω στις ερωτήσεις σας ε, για οποιασδήποτε λεπτομέρειες που σχετίζονται με αυτές τις δραστηριότητες. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Βιεβουρόφσκι. Θα ακούσουμε τώρα τον καθηγητή Πελεγκρινή που είναι ο πρόεδρος του Συμβουλίου Συνεργασίας της Ευρωπόλ. Και εσείς έχετε 12 περίπου λεπτά, ελαστικός χρόνος, αλλά θα αφήσουμε και λίγο χρόνο για υποβολή ερωτήσεων και χωρίς απαντήσεων. Αλλά μπορείτε να ζητήσετε ήδη από τώρα το λόγο γραπτός. Έχετε το λόγο κύριε Πελεγκρίνη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητά μέλη του Ευρωπαϊκού και των Εθνικών Κοινοβουλίων, αξιότιμοι αξιωματούχοι, Ω πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, του Συμβουλίου Συνεργασία Ευρωπόλ, χαίρομαι ιδιαίτερω για την τιμή που μου δίνετε να σα ενημερώσω για τι πρόσφατε δράσει και προοπτικέ του Συμβουλίου Συνεργασία τη Ευρωπόλ. Ε, Συνεχίζοντα την πρώτη ενημέρωση που σα έκανα πέρυσι το Φεβρουάριο στο Βουκουρέστι. Όπω ξέρετε, από την θέση ισχύ του κανονισμού της, Ευρωπόλ, ο, Ευρωπαϊκός, ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων είναι ο επόπτης όλων των δραστηριοτήτων επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων των κοινωτικών θεσμικών οργάνων και οργανισμών και είναι τώρα η αρμόδια αρχή για τον έλεγχο νομιμότητα επεξεργασία δεδομένων που πραγματοποιεί και η Ευρωπόλ. Βέβαια, η συμμετοχή των εθνικών αρχών προστασία δεδομένων είναι σημαντική γιατί η μεγάλη πλειοψηφία των δεδομένων που συγκεντρώνει και επεξεργάζεται η Ευρωπόλ προέρχονται από τα κράτη-μέλη και σε κάποιο βαθμό επιστρέφουν ή επιστρέφονται και στα κράτη-μέλη αυτά τα δεδομένα. Για το λόγο αυτό το άρθρο 45 του κανονισμού για την Ευρωπόλ, για τον Ευρωπόλ μάλλον, έχει θεσπίσει το ε, Συμβούλιο Συνεργασίας ε, τη Ευρωπόλ που απαρτίζεται από τον Ευρωπαίο Επόπτη και τι Εθνικέ Εποπτικές αρχέ. και η επικοδομητική του συνεργασία προβλέπεται στα άρθρα 44 και 45 του κανονισμού τη Ευρωπόλ και επιτρέπει συντονισμένη εποπτεία όλων των ροδεδομένων που κατευθύνονται προς την Ευρωπόλ και εκπορεύονται από αυτήν, κάτι που είναι απαραίτητο για να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις, ε, τις επεξεργασίες των δεδομένων με τις ειδικέ ε, διατάξεις που προβλέπεται στην Ενωσιακή Νομοθεσία. Στην επιχειρησιακή πλευρά διαθέτουμε μία ομάδα εθνικών εμπειρογνωμόνων που συμμετέχουν σε όλες τις επιθεωρήσεις ε, της Ευρωπόλ που οργανώνονται από τον Ευρωπαίο Επόπτη. Και αυτή η επιχειρησιακή συνεργασία ε, στόχο έχει να διατηρηθεί ένα υψηλό επίπεδο γνώση ό,τι αφορά τη λειτουργία τη Ευρωπόλ ε, και να εξοικειωθούν με τον έλεγχο αυτό όλε οι εθνικές εποπτικέ αρχές. Και έτσι βοηθούνται και οι εποπτικέ αρχές να διεξάγουν τους δικέ του επιθεωρήσει σε εθνικό επίπεδο και συμμετέχουν σε ένα πανευρωπαϊκό δίκτυο πραγματογνωσύνη και επαγγελματικών σχέσεων που τροφοδοτεί την κοινότητα αυτή. Ε, εμείς ε, συναντιόμαστε δύο φορές το χρόνο και η τελευταία συνάντηση έγινε το 2019. Τότε το Συμβούλιο Συνεργασίας υιοθέτησε την έκθεση δραστηριοτήτων, το πρόγραμμα δραστηριοτήτων για τη διετία 2018-2020 και ενημέρωσε το πρόγραμμα εργασιών επίση για το 2018-2020. Θα δείτε σε αυτά τα δύο έγγραφα την εκθεση περγαμενο πεπεργαμένο 17-18 και το πρόγραμμα εργασιών για το 18-20 τι δραστηριότητε μα στο παρελθόν, παρόν και μέλλον. Πρόσφατα το Συμβούλιο Συνεργασία εκπόνησε γνωμοδοτήσει για δύο συναφή θέματα. Το Φεβρουάριο του 2019 εκπονήσαμε τη γνωμοδότηση για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Παρακολούθηση Εντοπισμού, το σχέδιο που προειδοποιεί για κινδύνους παράνομης διασυνοριακής ανταλλαγής δεδομένων για εντοπισμού. Εκεί συστήσαμε στους συνομοθέτες ε, να προτείνουν κατεπηγόντως τη δημιουργία της κατάλληλης νομικής βάσης τον τρέχοντα μήνα στείλαμε στον πρόεδρο του, του δικτύου μονάδων χρηματοοικονομικών πληροφοριών, του FUNET, την γνώμη ότι το FUNET δεν μπορεί να υποφεληθεί από την τεχνική ε, υποδομή για την ανταλλαγή επιχειρησιακών δεδομένων, γιατί οι κατηγορίες των υποανταλλαγή δεδομένων δεν συνάδουν με την εντολή της Ευρωπόλ. Και στις δύο περιπτώσεις ανακύπτει ανάγκη εξασφάλισης των κατάλληλων νομικών βάσεων και των επιχειρησιακών μέσων για την απεξεργασία των δεδομένων ώστε να εξασφαλίσουμε και την αποτελεσματικότητα και τη σωστή ε, εφαρμογή του νόμου ε, με ταυτόχρονο σεβασμό των προσωπικών δεδομένων που τη χάνουν επεξεργασία. Και από αυτή την άποψη είναι σημαντικό και στη μελλοντική επεξεργασία αλλά και στα μελλοντικά καθήκοντα, τα επιπλέον καθήκοντα της Ευρωπόλ να τηρήσουμε την εντολή και το νομικό πλαίσιο που έχουν αποφασίσει και θεσπίσει οι συνομοθέτες. Οποιαδήποτε επεξεργασία που υπερβαίνει την παρούσα εντολή θα πρέπει να ορίζετε να οριθετείται αυστηρά από τον νόμο. Το, θέμα του τη κατάλληλη εντολή και της εποπτείας δεν περιορίζεται στις περιπτώσει αυτέ. Πολλά νέα ε, συστήματα πληροφόρησης και επιχειρησιακοί φάκελοι έχουν προβλεφθεί, όπως το ΕΤΙΑ, το Ευρωπαϊκό ε, Σύστημα Πληροφοριών Ταξιδιού και Διοδότησης, ή το Σύστημα Εσόδου-Εξόδου. Επίσης υπάρχει ήδη η όθηση υπέρ αυτής της διασύν, διασύνδεσης που εσφαλμένα αποκαλείται διαλειτουργικότητα για πολλά από τα θέματα αυτά, καθώς και το σύστημα πληροφοριών της Ευρωπόλ, το EIS. Από αυτή την άποψη η διασύνδεση είναι από μόνη της μια επεξεργασία που χρήζει εποπτείας, προκειμένου να εξασφαλιστεί η αναλογικότητά της και η εφαρμογή των ε, ατομικών θεμελιωδών δικαιωμάτων. Ένα από τα βασικά μέσα του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων είναι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων που έχει λάβει νομική προσωπικότητα και στόχο έχει την ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού δόγματος προστασίας δεδομένων με υψηλό επίπεδο συνεργασίας και συνοχής ε, μεταξύ των ενδιαφερομένων. Με βάση το νέο αυτό πλαίσιο, οι αρμόδιοι για την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι νομοθέτες, έχουν καθορίσει ένα τρόπο για συμπερίληψη των ad hoc ε, ομάδων συντονισμού εποπτείας μαζί με, ε, με το σύστημα, Schengen, σύστημα πληροφοριών Schengen, το σύστημα πληροφοριών των τελωνίων και το σύστημα ενημέρωσης για τις θεωρήσεις και να τις συμπεριλάβει αυτά σε ένα ε, συνεκτικό πλαίσιο. Και μάλιστα με την αναδιατύπωση του κανονισμού 45-2001 έχουμε ε, συζήτηση ε, της γενικής εποπτείας που ασκεί το Ευρωπαϊκό Σύμβουλιο Προστασίας των Δεδομένων προκειμένου να υπερκεραστούν οι κατακαιρματισμοί ε, της προηγούμενης νομοθεσίας. Και μάλιστα αυτό το νέο μοντέλο συντονισμένης εποπτείας θα καθιερωθεί επίσημα από το Συμβούλιο Προστασία Δεδομένων στα τέλη του έτου. Το Συμβούλιο συνεργασία τη Ευρωπόλ κρίνει θετικά τη συμπερίληψή του στο μέλλον της διαδικασία, στη διαδικασία αυτή, γιατί θα συνάδει στη συνοχή και τη συνεκτικότητα των υποπτικών δραστηριοτήτων των συστημάτων πληροφοριών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και μάλιστα μια τροπολογία στον κανονισμό της Ευρωπόλ θα καταστεί αναγκαία προκειμένου να ε, ε, γίνει πραγματικότητα αυτή η συμπερίληψη. Αυτό θα γίνει εν ευθέτω χρόνο, το, το νέο μοντέλο γίνει πλήρω λειτουργικό. Γιατί ε, προτεραιότητά μας είναι μια ε, ομαλή και αποτελεσματική υλοποίηση των αποστολών μας. μία, από τις αποστολές μα, μία από τις αποστολές μας είναι η προστασία των δεδομένων ε, να είναι πιο αποτελεσματική. είναι σημαντικό να γίνεται επικαιροποίηση των δεδομένων ε, και κυρίως να ενημερώνεται καλύτερα το κοινό, όπως στα φυλάδια ε, γνώρισε τα δικαιώματά τους. Από αυτή την άποψη, ε, μερικές φορές ο κόσμος βρίσκεται ανήμπορος και χαμένος μπροστά στην πολυπλοκότητα των διατάξεων. Γι' αυτό και είναι σημαντικό οι ομάδες συντονισμού εποπτείας να εξασφαλίσουν καλύτερη πρόσβαση και όλες οι διαθέσιμες πληροφορίες να δίνονται στο κοινό προκειμένου να διευκολυνθεί η εποπτεία των δεδομένων άσχετα από το σύστημα που εφαρμόζεται. Και το Συμβούλιο Συνεργασίας πολύ ευχαρίστω ε, θα συμμετάσχει σε αυτή τη διαδικασία σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ε, κάτι που είναι σημαντικό ε, και με τη συμμετοχή του επόπτη προστασία δεδομένων. Ένα άλλο σημαντικό θέμα αφορά την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ της Ευρωπόλ και, των τρίτων, και χωρών. Μέχρι στιγμής η Ευρωπόλ είναι συμβαλόμενο μέρος σε διάφορες συνεργασίες, ε, συμφωνίες ε, επιχειρησιακής συνεργασίας που, που περιλαμβάνουν ανταλλαγή προσωπικών δεδομένων με 8 τρίτε χώρε. Αλβανία, Αυστραλία, Βοσνία, Ερζεγοβίνη, Καναδάς, Κολομβία, Γεωργία, Ισλανδία, Λίχτενστάιν, Μολδαβία, Μονακό, Μαυροβούνιο και Βόρεια Μακεδονία. Το άρθρο 25, παράγραφος 4 του κανονισμού τη Ευρωπόλ προβλέπει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να επανεξετάσει όλες τις συμφωνίες συνεργασίας που συνήψε στο παρελθόν με τρίτες χώρες και αυτό μέχρι το 2021. Παρόλο που όλες αυτές οι χώρες διαθέτουν νομοθεσία για την προστασία δεδομένων και πάνω κάτω ε, διαθέτουν και ανεξάρτητες αρχές προστασίας δεδομένων, είναι σημαντικό να γίνει επανεξέταση και επαναθεώρηση αυτών των συμφωνιών το συντομότερο δυνατό για πολλούς και διάφορους λόγους. Καταρχάς, η ανταλλαγή προσωπικών δεδομένων με τις χώρες αυτές δεν θα πρέπει να διακοπεί μετά την προθεσμία αυτή. Ε, ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να τηρείται το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προστασίας Δεδομένων. Δεύτερον, στις 20 Δεκεμβρίου του 2017 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε οκτώ συστάσεις ε, για αποφάσεις του Συμβουλίου προκειμένου να επιτρέπει την έναρξη διεθνών διαπραγματεύσεων για σύναψη διεθνών συμφωνιών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οκτώ χωρών της Μέσης Ανατολής και Βορείου Αφρικής την Αλγερία, το Αίγυπτο, την Αίγυπτο, το Ισραήλ, η Ορδανία, Λίβανο, Μαρόκο, την Ισία και Τουρκία. Τέτοιες διεθνείς συμφωνίες ε, θα παρέχουν την κατάλληλη νομική βάση για την ανταλλαγή προσωπικών δεδομένων μεταξύ Ευρωπόλ και αρμόδιων αρχών των τρίτων χωρών, ε, των αρχών αρμόδιων για την καταπολέμηση σοβαρών εγκλημάτων και τρομοκρατίας. Επίσης, στις 4 Ιουνίου του 2018, το Συμβούλιο υιοθέτησε τις αποφάσεις που επιτρέπουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με όλες αυτές τις τρίτες χώρες. Και μάλιστα το Συμβούλιο Συνεργασίας θεωρεί ότι αυτές οι περιπτώσεις είναι καλή ευκαιρία για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καθορίσει ένα γενικότερο πλαίσιο συμφωνιών με βάση ε, τις προδιαγραφές προστασίας δεδομένων που θέτει η Οδηγία του 2016-680. Και αυτό το πλαίσιο γενικής εφαρμογής θα καθορίζει μηχανισμούς για την έμπρακτη παρακολούθηση των μεμονωμένων συμφωνιών και θα περιλαμβάνει και περιοδικούς ελέγχους και αξιολογήσεις και επιτόπιες επιθεωρήσεις προκειμένου να αξιολογηθεί η λειτουργία του σε σχέση με τις επιχειρησιακές ανάγκες Ευρωπόλ καθώς και η προστασία των ευρωπαϊκών αρχών και δικαιωμάτων και προστασία των δεδομένων. Και μάλιστα, όπως φαίνεται στην επιστολή της 19 Αυγούστου του 2019 προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβούλιο Συνεργασίας Ευρωπόλ έχει δεσμευθεί πλήρως να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυ στην διαδικασία αναθεώρησης και να συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε αυτή τη σημαντική δραστηριότητα. Θα ήθελα, όπω και στην προηγούμενη μου ενημέρωση, να τονίσω το γεγονός ότι το Συμβούλιο Συνεργασίας της Ευρωπόλ είναι υπέρ μιας ανοιχτής και διαφανούς εφαρμογής ε, της αποστολής του, προκειμένου το πλαίσιο προστασίας δεδομένων της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης να γίνει πραγματικότητα και για τον οργανισμό και για τους πολίτες. Και χαιρετίζουμε την εποπτεία της ΜΟΚΕ σε αυτά τα σημαντικά θέματα και σας διαβεβαιώ για την προθυμία μου να σας ε, ενημερώσω και να σας παράσχω όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε. Ευχαριστώ. Thank you. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα θα ακούσουμε τους συναδέλφους. Δύο λεπτά ο χρόνος ομιλίας και στο τέλος θα δώσουμε και πάλι τον λόγο στον κύριο Βιβορόφσκι και τον καθηγητή τον κύριο Πελεγκρινή. Κύριος το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχω κάποιες ερωτήσεις στον βοηθό επόπτη προσωπικών δεδομένων. Το ένα αφορά το θέμα της διατήρησης των δεδομένων, ένα από τα πιο δύσκολα ζητήματα της ε, παρακολούθησης γιατί αφορά τις καθημερινές μας επικοινωνίες και κινήσεις. Η Europol ε, είναι υπέρ της επανεισαγωγής ε, μιας τέτοιας πολιτικής υπό το όνομα της περιορισμένης διατήρησης των δεδομένων, δηλαδή να εξαιρούνται κάποιοι επαγγελματίε, αλλά κατά τα άλλα καλύπτεται όλος ο πληθυσμός. Παραδείγματος χάρη είχαν φιλοξενήσει ένα εργαστήριο για το θέμα αυτό και έχετε εμπλακεί εσείς καθόλου σε αυτήν την διαδικασία υπό την ιδιότητά σας και συμφωνείτε ότι το να εξαιρούνται κάποιοι επαγγελματίες δεν πληρεί τα κριτήρια του ε, ΔΕΚ, το οποίο λέει ότι πρέπει να υπάρχει μία σχέση μεταξύ του κάθε ατόμου του οποίου τα δεδομένα διατηρούνται και, ένα, και ενός σοβαρού εγκλήματος. Το δεύτερο μου ερώτημα αφορά ε, την ε, συμφωνία SWIFT ε, που αναφέρατε και το ζήτημα χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Έχει επισημανθεί ότι οι ΙΠΑ βασικά αποθηκεύουν τα δεδομένα βάσει αυτής της συμφωνίας για πάντα, γιατί οι αρχές δεν λένε πότε ολοκληρώνονται οι έρευνες. Οπότε, τι προτείνετε εσείς να γίνει για αυτό και γιατί η Κομισιόν συμπεραίνει ότι ε, κατά βάση όλα αυτά είναι ε, συμβατά με την συμφωνία. κυρία Αμιτάκα από την Γερμανία έχετε τον λόγο. Ευχαριστούμε πολύ που μου δίνετε τον λόγο. Όταν μιλάμε για τον έλεγχο όλων των συμφωνιών μέχρι το 2020 με τις τρίτες χώρες, ε, θέλω να σας ρωτήσω από την πρώτη ενδεκάτου τι θα γίνεται με τα δεδομένα με την, που ανταλλάσσουμε με, την με το Ηνωμένο Βασίλειο. Δεν υπάρχει κάποια συμφωνία αυτή τη στιγμή. Μόλις θα γίνει η τρίτη χώρα, θα να κανείς ότι θα υπάρχει κάποιο είδους ε, συμφωνία η οποία θα συναυθεί με κάποιο τρόπο απόψη προστασία δεδομένων. Λοιπόν, τι θα γίνει αν δεν υπάρχει συμφωνία από την πρώτη δεκάτου And Then... Σα ευχαριστώ. Πάρα πολύ, κυρία Κινίτση, Ευρωβουλευτή, έχετε τον λόγο. Ναι, ευχαριστώ, κύρια Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα να κάνω μια προσωπική παρατήρηση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον πρόεδρο Λόπεζ Αγγιλάρ και θα ήθελα να υπενθυμίσω σε αυτή την φάση τον Τζάνι Μπουταρέλη και εγώ με την σειρά μου ένα προσωπικό μου φίλο ο οποίος πραγματικά έδωσε μια μεγάλη όθηση στην δραστηριότητα αυτή του EDPS και γι' αυτό τον ευχαριστώ. Ε, ευχαριστήσω και τους ε, καλεσμένους μας, οι οποίοι ανέφεραν βεβαίως τα της ε, δουλειάς τους. Τώρα, έχω μία ερώτηση η οποία αναφέρεται στο ViewNet. Το ViewNet είναι ένα αποκεντρωμένο δίκτυο, το είπαμε, το οποίο διαχειρίζεται η Europol, το οποίο συνενώνει τις διάφορες μονάδες ε, οικονομικών πληροφοριών. Υπάρχει η οδηγία αυτή του 2019 για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των διοκτικών αρχών και είναι ένα από τα πιο σημαντικά τεχνικά μέσα μέσω του οποίου γίνεται ανταλλαγή ε, πληροφοριών ε, Παραλύλουμε με το σύστημα Λοιπόν, υπό το φως ας πούμε των συστάσεων που έκανε η Europol θα ήθελα εγώ να γνωρίζω ποιες αλλαγές, ποιες βελτιώσεις μπορούν να γίνουν στο ViewNet έτσι ώστε να ενισχυθεί κυρίως ε, όσον αφορά όπως είπαμε την προοπτική αυτή της οδηγίας του 2019 δεδομένης της σημασίας που έχουν ε, οι συναλλαγές αυτές ε, σε σχέση με τα διασυνοριακά εγκλήματα. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και εγώ. Η κυρία Ντέιλι, Ευρωβουλευτής, σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, είμαι νέα σε αυτήν την Επιτροπή, οπότε προσπαθώ λίγο να δω την σχέση μεταξύ Europol και επόπτη προσωπικών δεδομένων. Εάν δούμε παραδείγματος χάρη το σύστημα πληροφοριών της Europol και πούμε ότι η επεξεργασία δεδομένων για μετανάστες στα hotspot που έχει εξετάσει ο επόπτης τα τελευταία χρόνια. Πώς γίνεται τελικά, από ό,τι αντιλαμβάνομαι η Frontex ε, παίρνει συνέντευξη από κάποιον, εάν διαπιστώσει κίνδυνο ζητείτε από την Interpol να κάνει κάποιον έλεγχο. Τι έλεγχο λοιπόν κάνετε εσείς, ε, μιλάμε για ε, δακτυλοσκόπηση, έλεγχο δεδομένων, διαβούλευση με τρίτη χώρα. Εάν υπάρχει διαβούλευση με τρίτη χώρα, πώς προσπαθούμε να προφυλαχθούμε από το ότι κάποιος παραδείγματο χάρη διαφεύγει λόγω πολιτικών διώξεων προφανώς η χώρα του δεν θα μας δώσει θετικές ας πούμε πληροφορίες τι γίνεται αν ο αξιωματικός Europol επισημάνει κάποιον ως κίνδυνο ασφαλείας και τι ε, μπορεί να κάνει αυτό το άτομο ως αντίδραση και αν έχετε κάποιο πρόβλημα εσείς ε, με αυτές τις ε, διευθετήσεις, αν έχουν υπάρξει κάποιε αλλαγέ και στο πλαίσιο αυτό και στο πλαίσιο των άλλων έρευνων του επόπτη ποιες διορθωτικές, ε, μάλλον υπήρξαν διορθωτικές ε, δράσει στι περισσότερε περιπτώσει, θεωρείται ότι συμμορφώθηκαν ή ε, υπήρχαν περιπτώσεις οποίε δεν χρειάστηκε γιατί εγώ αντιλαμβάνομαι για αυτά τα οποία λέτε για το πρόγραμμα χρηματοδότηση τη τρομοκρατία θα δημοσιευτεί, θα δημοσιευτεί όλο ή θα δημοσιευτούν μόνο μέρη του. Και επίσης αν μπορείτε να μας εξηγήσετε, ξέρω πως υπήρχαν λίγα παράπονα, ε, ποιες προσφυγές δεν έγιναν δεκτές όμως. Αν μπορείτε να μας δώσετε μία ιδέα. Σας ευχαριστώ. Θα δώσω τον λόγο τώρα στον κύριο Ριαμπόφσκι. Σας ευχαριστώ. Να απαντήσω λοιπόν στις ερωτήσεις ε, που έγιναν. Ξεκινάμε από το θέμα της διατήρησης των δεδομένων. Ξέρω πως ε, έχετε κάνει την ίδια ερώτηση και στην ε, συνειδρίαση της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ με την Europol. Οφείλω να πω ότι έχω μια διαφορετική άποψη από εσάς όσον αφορά την γενική πιο γενικό σκεπτικό της υποχρεωτικής ε, διατήρησης δεδομένων και τις άλλες πτυχές. Αυτό το οποίο μπορώ να πω εγώ από τη δικιά μας τη σκοπιά του επόπτη, γιατί δεν μπορώ να σας πω την άποψη της Europol, είναι ότι ε, είμαστε σίγουροι βεβαίως ότι η διακράτηση αυτή υπάρχει ως διαδικασία. Το θέμα είναι κατά πόσον είναι υποχρεωτικό το σύστημα και το σημαντικότερο είναι το δικαίωμα πρόσβασης σε αυτά τα δεδομένα. Ποιος έχει δικαίωμα πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα, ποια θεσμικά όργανα, ποιες υπηρεσίες, για ποιο λόγο και για ποιες ε, έρευνες. Υπάρχει η δυνατότητα έρευνας ε, των δεδομένων για να βρεθούν ε, εγκληματικέ δραστηριότητες ή απλά αναζητούν πράγματα τα οποία είναι τώρα υπό έρευνα. Γνωρίζετε επίσης ε, και οι περισσότεροι νομίζω που είναι στην Ελλάδα γνωρίζουν ότι ε, παράλληλα υπήρχε και η συζήτηση στο ΔΕΚ, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και ε, είχαμε την εκδίκαση, συνεκδίκαση τεσσάρων υποθέσεων από διάφορες οργανώσεις που αμφισβητούσαν την διαδικασία και αναμένουμε την απόφαση του 10. Αυτή τη στιγμή μπορώ να πω ότι δεν υπάρχει κάποια διαδικασία ενιαία διακράτηση των δεδομένων. Υπάρχουν διαφορές μεταξύ ε, των χωρών, κάτι το οποίο ακριβώς καταλήγει στις ε, διαφορές ε, στα δεδομένα που αποστέλλονται στην Europol ε, τελείως διαφορετικά τηλεπικοινωνιακά δεδομένα και με τα μεταδεδομένα του διαδικτύου. Και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι κομμάτι της δραστηριότητάς μας, ειδικά της εποπτικής. Όσον αφορά το SWIFT ε, τώρα και τα όσα συνδέονται με την παρακολούθηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας γνωρίζουμε τον πολύ περιορισμένο αντίκτυπο που έχει η Europol στις ε, καθημερινές δραστηριότητες ε, των ε, θεσμικών οργάνων που καλύπτονται από αυτή την συμφωνία και οπωσδήποτε αυτό θα πρέπει να αποτελέσει τμήμα της επανεξέτασης αυτής της διαδικασίας που αυτή τη στιγμή γίνεται αφού έχουν εισαχθεί οι νέοι κανονισμοί και ο κανονισμός για την προστασία των δεμένων. Η έκθεση ε, θα δημοσιευτεί ολόκληρη μετά την ε, επιθεώρηση. Μία σύσταση υπάρχει, η οποία είναι τεχνικής ε, φύσεως. Υπάρχουν λοιπόν 8 συστάσεις, 7 θα είναι δημόσιες και το υπόλοιπο έγγραφο θα είναι επίσης δημόσιο. Οπότε αποφασίσαμε ότι το έγγραφο αυτό πρέπει οπωσδήποτε να είναι δημόσιο. Για το Brexit. Ε, το Brexit ε, δημιουργεί τα προβλήματα τα οποία βεβαίως εν μέρη θα λυθούν με την συμφωνία εάν υπάρξει συμφωνία. Η πιο δύσκολη κατάσταση θα είναι εάν έχουμε το λεγόμενο σκληρό Brexit και θα πρέπει κάποια μέρα να δούμε τις μεγάλες αλλαγές στη συνεργασία με το Ηνωμένο Βασίλειο. Έχουμε αρχίσει να εξετάζουμε δύο λύσεις. Ταυτόχρονα η πρώτη είναι μια λύση που θα λέει το τι θα συμβεί στις 31 Οκτωβρίου, ποια δεδομένα μπορούν να παραμείνουν στην Europol και ποια μπορούν να δοθούν και υπό ποιες συνθήκες στο Ηνωμένο Βασίλειο και αυτό είναι το έγγραφο το οποίο ακόμα συντάσσεται αλλά βεβαίω, είμαστε σίγουροι ότι θα εγκριθεί από την Europol και το Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την ημερομηνία αυτή και η γενική μας ανησυχία είναι ακριβώς ε, η συνεργασία μεταξύ των διοκτικών αρχών και της Europol που θα πρέπει να είναι τουλάχιστον επιχειρησιακή και αποτελεσματική μετά από αυτό έχοντας κατά νου ότι την πρώτη μέρα δεν θα έχουμε επίσημη συμφωνία μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Ευρωπαϊκής Ένωσης για το μέλλον αυτής της συνεργασίας. Οπότε αυτό το εξετάζουμε. Ταυτόχρονα συζητούμε για την πιθανότητα να εφαρμόσουμε κάποια μοντέλα παρόμοιας συνεργασίας όπου έχουμε επιστροφή δεδομένων σε τρίτες χώρες. Αυτό βέβαια σχετίζεται και με τη συζήτηση ε, για τις 8 χώρες με τις οποίες το Συμβούλιο θα εξετάσει πιθανότητα ανταλλαγής δεδομένων. Ε, πρόκειται κυρίως για χώρες της ε, Μέσης Ανατολής και Βορείου Αφρικής, αλλά δεν έχουμε ακόμη πληροφορίες για, το, για την αλλαγή αυτής της συνεργασίας. Είναι θέμα που αφορά τους εκπροσώπους ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ξεκίνησαν τις διαπραγματεύσεις με τις τρίτες αυτές χώρες. Ό,τι αφορά το FIUNET, ε, το δίκτυο για των μονάδων, ομάδων, των ομάδων, του μονάδων χρηματοοικονομικής πληροφορίας, οι επιχειρήσεις που γίνονται σε αυτό το FIUNET, FIUNET περιλαμβάνουν δεδομένα περισσότερα από αυτά που μπορεί να συγκεντρώσει και να επεξεργαστεί η Ευρωπόλ. Δηλαδή ξεπερνούν ε, την εντολή ε, της Ευρωπόλ. Και αυτό είναι κρίμα πραγματικά, γιατί το FUNET θα ήταν ένα πολύ αποτελεσματικό τρόπο συνεργασία. Αλλά απ' την άλλη, η νομιμότητα είναι η παριθμόν ένα προτεραιότητα και το παριθμόν ένα ζητούμενο. Ή, πολλό δε μάλλον που μιλούμε για τι ε, αρχέ επιβολή του νόμου και για τη δυνατότητα ανταλλαγή τέτοιων δεδομένων από αυτέ. Ευχαριστώ. συνεχίστε εσείς. Εδώ βλέπετε την ε, ε, πολύ ε, αγαστή συνεργασία μεταξύ του ΕΠΟΠΤΗ και των Εθνικών Αρχών. Να συνεχίσω την ερώτηση για το FIUNET. Το δίκτυο μονάδων χρηματοοικονομικών πληροφοριών είναι αποκεντρωμένο και τη διαχείριση την εξασφαλίζουν τα ίδια τα κράτη-μέλη μάλιστα από νομικής πλευράς ε, στηρίζεται σε διμερείς συμφωνίες μεταξύ των χωρών για ανταλλαγή πληροφοριών. Οπότε η τεχνική υποδομή που επελέχθη τότε για το FUNET ανταποκρινόταν στο μοντέλο αυτό και στηριζόταν σε ανταλλαγές μεταξύ ισοτήμων. Το πρόβλημα που ανακύπτει τώρα και οφείλεται στην επιτυχία του FUNET είναι ότι η τεχνική υποδομή που το χαρακτηρίζει δεν μπορεί να αναβαθμιστεί, γιατί είναι πολύ μεγάλος όγκος πληροφοριών που ανταλλάσσουν τα μέλη του FUNET. Και γι' αυτό υπάρχουν κίνητρα για την παρέμβαση της Ευρωπόλ, που θα είναι ένας τεχνικός πάροχος και θα συγκεντρώνει τα τεχνικά μέσα σε ένα κεντρικό επίπεδο, με βάση το συστημα ανταλλαγη ανταλλαγής μηνυμάτων C1, χωρίς όμως να τροποποιεί το τη νομική διάρθρωση, τη νομική δομή του συστήματος. Και όπως είπε ο κ. Βεβουρόφσκι, υπάρχουν κάποια θέματα που αφορούν το γεγονός ότι το FUNET κινητοποιείται από κάποια συστήματα κατώτατων των ορών. Αν μια συναλλαγή ξεπερνάει ένα κατώτατο όριο, τότε κινητοποιείται, ενεργοποιείται το σύστημα και κυκλοφορούν οι πληροφορίε στο σύστημα. Αυτέ όμω οι πληροφορίε εκφύσεω δεν συνδέονται με υπόπτου. Οπότε, ακόμη και πληροφορίε για μη υπόπτου κυκλοφορούν στο σύστημα. Και το ζήτημα που ανακύπτει, όπω αναφέρθηκε, είναι όταν εξετάζουμε την, Ευρωπόλ, την εντολή της Ευρωπόλη, η Ευρωπόλ μπορεί να διαχειριστεί μόνο πληροφορίες που αφορούν υπόπτους. Και όταν μιλούμε στο Συμβούλιο Συνεργασίας με τα κράτη-μέλη, σε κάποια ε, νομικά συστήματα, σε κάποια δικαϊκά συστήματα δεν υπάρχει καν νομικός ορισμός τι εστί ύποπτο. Οπότε αυτό δημιουργεί προβλήματα για τη νομική βάση που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη χρήση του συστήματος στην περίπτωση των υπόπτων, μια και μερικές χώρες δεν έχουν νομικό ορισμό για τον υπόπτο. Οπότε η απάντησή μου θα ήταν διπλή. Διτή. Δεν μπορούμε να έχουμε μια τεχνική λύση σε ένα νομικό πρόβλημα. Το πρόβλημα, το ζήτημα είναι, όπως είπα και στην ομιλία μου, είναι τι νομική βάση θα επιλεχθεί στο μέλλον για το FIUNET, για αυτό το δίκτυο μονάδο χρηματοοικονομικών πληροφοριών. Γιατί αν γίνει μια συγκέντρωση των πληροφοριών σε ένα κεντρικό σημείο. Δεν θα έχουμε πια συμφωνίες διακρατικές, αλλά θα έχουμε μια άλλη διαδικασία που θα απαιτεί και τον κατάλληλο έλεγχο και την κατάλληλη εποπτεία. Το πρόβλημα είναι ότι σήμερα δεν υπάρχει κατάλληλος μηχανισμός εποπτείας για το σύστημα αυτό ή για το μελλοντικό σύστημα όπως θα εξελιχθεί. Και αυτό θα πρέπει να ε, κατοχυρωθεί και νομικά και να οριοθετηθεί και νομικά. Οπότε, αν θέλουμε μια τεχνική αρρωγή που θα συνάδει με, την, με τα σημερινά χαρακτηριστικά του FIUNET, που είναι μεταξύ ομοτήμων, θα πρέπει να δούμε αν θα αναβάλουμε το πρόβλημα για το μέλλον ή θα εξετάσουμε αν η νομική δομή του συστήματος είναι δόκιμη, γιατί κάποιες χώρες θα πρέπει να επανεξετάσουν το καθεστώς των μονάδων του FIUNET και αυτό υπάρχει πρόβλημα, δημιουργεί πρόβλημα στον ορισμό του συστήματος, γιατί ένα σύστημα μεταξύ ομοτήμων έχει καθοριστεί ως, έχει επιλεγεί μάλλον ως λύση για να παρακαυθούν κάποια νομικά θέματα. Αυτό όμως δεν είναι αρκετό όταν θέλουμε ένα νομικό σύστημα ε, που θα είναι κεντρικό και θα συμπεριλαμβάνει και την Ευρωπόλ. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν από την αρχή το νομικό ζήτημα σε σχέση με το FUNET και το καθεστώς του. Για να απαντήσω εν συντομία στην ερώτηση για τα hot spot. θα έχουμε μια καλύτερη εικόνα της δομής ε, σε αυτό που θα σας στείλουμε γραπτός. Αλλά πρέπει να πω ότι τόσο η Ευρωπολ όσο και η Frontex συνεργάζονται με τις εθνικές αστυνομίες των κρατών μελών και η Ευρωπόλ εργάζεται βάσει του αιτήματο των εθνικών αρχών, ειδικότερα των εθνικών αστυνομικών αρχών. Τα κράτη-μέλη επίση έχουν απευθεία πρόσβαση στο ΙΕΣ και εάν οι έλεγχοι γίνονται σε αντιπαραβολή με τις βάσεις δεδομένων της Ευρωπόλ, ε, βασίζονται μόνο στα δεδομένα των υπόπτων, αλλά από ό,τι κατάλαβα η ερώτησή σα αφορούσε και τη συνεργασία με τρίτε χώρε και το ενδεχόμενο χρήση αυτού του αιτήματο με τρίτε χώρε. Αυτό, αν ε, δεν έχετε πρόβλημα, θα σα το στείλω γραπτό. Και το δεύτερο, οι ερωτήσει για τι καταγγελίε. Οι καταγγελίε που καταλήγουν στον NDPS αφορούσαν γενικώ την έλλειψη πρόσβαση στα δεδομένα που αποθηκεύει η Ευρωπόλ. Οπότε Απλά μιλάμε για περιπτώσεις όπου δεν δόθηκαν σωστέ πληροφορίε στους ανθρώπου για τα δεδομένα του κατά πόσο είναι αποθηκευμένα ή όχι στην Ευρωπόλ. Αλλά όπως είπα, από τις καταγγελίες που έχουμε λάβει, οι μισές ουσιαστικά δεν είναι παραδεκτές, διότι δεν εστάλησαν στο σωστό ε, αποδέκτη. Αγαπητέ καθηγητά Πελεγκρίνη, αγαπητέ κύριε Βιβιερόφσκι, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και τους δύο πολύ και για τις δύο παρουσιάσεις σας. Ευχαριστώ και τους συναδέλφους για τις πολύ καλές ερωτήσεις. Χουάν, λοιπόν, έχουμε περάσει 4,5 σχεδόν ώρες ε, συνεχής συζήτησης. Ελπίζω να ήταν επικοδομητικές για όλους μας. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη συμβολή σας, την συνεργασία σας, την παρουσία σας και την προσοχή σας. Δεν έχω παρά να σας υπενθυμίσω ότι έχετε πρόσκληθει στη δεξίωση που θα έχουμε απόψε στον, Ευρωπαϊκό, στον οίκο της Ευρωπαϊκής Ιστορίας. Λίγα μέτρα από εδώ, αλλά για όσους από εσάς δεν γνωρίζετε την περιοχή εδώ των Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων, να σας ανακοινώσω ότι θα υπάρξουν υπάλληλοι, μέλη του προσωπικού που θα σας καθοδηγήσουν μέχρι τον οίκο Ευρωπαϊκής Ιστορίας. Η δεξίωση θα αποτελέσει μια ευκαιρία να συνεχίσουμε τη συζήτηση που κάνουμε σήμερα σε ένα πιο άτυπο χώρο. Και ως κύριο μιλητή θα έχουμε τον Επίτροπο για την Ασφάλεια, τον Julian King ο οποίος ε, θα εκφωνήσει μια σύντομη ομιλία ε, επ' ευκαιρία αυτής της ε, εκδήλωσης και θα συνεχίσουμε τις εργασίες μας αύριο στις 9 το πρωί στην ίδια αίθουσα. Παρακαλώ λοιπόν, κρατήστε τις κονκάρτες που σας δόθηκαν που σας επιτρέπουν την ταυτοποίηση και την είσοδο τόσο στο Νίκο Ιστορίας όσο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αύριο το πρωί στις 9 το πρωί στην ίδια αίθουσα. Ευχαριστώ πολύ, θα τα πούμε σε λίγο.